Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι ένας ε, Ιταλός στρατιωτικός ε, έχασε την ζωή του σε μία ανταλλαγή πυρών ε, στο Αφγανιστάν. Πρόκειται για τον Λούκα Σάνα, στην οικογένεια του οποίου αποστέλουμε τα συλληπιτήριά μας. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη λοιπόν αφορά την δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση στην ΑΙΤ ένα χρόνο μετά από τον σεισμό. Συγκεκριμένα ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση. Δίνω αμέσως το λόγο ε, εξ ονόματος της Επιτροπής ε, στην Επίτροπο κυρία Γεωργίευα. Παρακαλώ. Thank you, Madam President. And may I also join you in expressing sympathy. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με την ε, σειρά μου να αποστείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια όσων έχασαν τη ζωή τους. Ο σεισμός στην Αιτία ένα χρόνο πριν αποτελεί μία από τις ε, σοβαρότερες φυσικές καταστροφές που συνέβησαν στον πλανήτη μας τα τελευταία χρόνια. Αλλά αποτέλεσε ε, και μία βέλτιστη ευκαιρία για την επίδειξη αλληλεγγύης και ανθρωπισμού. Επίσης ε, ήταν μια ευκαιρία για να μάθουμε όλοι μας ένα μάθημα κουράγιου και θάρρους. Βεβαίω, πρώτα απ' όλα θέλουμε να ε, στείλουμε τη σκέψη μας σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και σε όσους επέζησαν ε, και που επέζησαν και λόγω της ε, δικής μας στάσης πρέπει να σας πω ότι εμείς κινητοποιήσαμε όλες τις διαθέσιμες ενέργειες και πράξεις έτσι ώστε να δώσουμε ε, όσο γίνεται περισσότερη ε, ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και αναπτυξιακή βοήθεια όπως σας αναφέρει αργότερα ο Επίτροπος Πίμπολς. Δώσαμε 130 30 ε, εκατομμύρια μόνο σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανθρωπιστική βοήθεια και βεβαίως πολύ περισσότερα χρήματα ε, εστάλησαν στην IT. Ε, 4 εκατομμύρια ανθρώπους περιθάλψαμε. 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι βρήκαν στέγη και έτσι ώστε να μπορέσουν να ξαναξεκινήσουν τη ζωή, ζωή τους η βοήθειά μας δεν αφόρασε μονάχα το Πόρτο ε, Πρένς, αλλά και άλλες ε, περιοχές που είχαν ε, θυγεί και βοηθήσαμε επίσης και 500.000 Αιτινούς να εγκαταλείψουν την πόλη του Πόρο Πρένς και να, πούν, να πάνε κοντά σε, στην οικογένειά τους όπου θα μπορούσαν να επιβιώσουν η παρούσα ανθρωπιστική βοήθεια ε, αφορά 22 εκατομμύρια τα οποία ε, ε, προσπαθούν να καλύψουν βασικές ανάγκες επιδημιολογικές έρευνες, αναλώσιμα, εκπαίδευση. Έχουμε δώσει καθαρό νερό σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους και έχουμε Έχουμε επίσης ε, ε, βοηθήσει πάρα πολλούς ε, ανθρώπους να ξεπεράσουν τη χολέρα και να μάθουν πώς μπορούν να προφυλακτούν από την χολέρα μέσω μαθημάτων προς την κοινότητα. Ε, ελπίζαμε ότι ένα χρόνο μετά από το σεισμό θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Ε, αυτή τη στιγμή όμως δυστυχώς δεν μπορούμε να το πούμε. Ε, ακόμα δίνουμε 33 εκατομμύρια για το 2011 με εστίαση κυρίως στην περίθαλψη την υγειονομική φροντίδα. Βεβαίως εξακολουθούμε να προσπαθούμε τα μέγιστα όσον αφορά την υγιεινή, γιατί βεβαίως αποτελεί ένα μέγιστο κίνδυνο για επιδημίες, άρα μεγάλο κίνδυνο για τον ε, πληθυσμό. Ε, ε, ξέρετε ότι το σύστημα υγείας της ΑΙΤΙΣ έχει εντελώς καταστραφεί, άρα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να το ξαναφτιάξουμε. Έχουμε βασιστεί σε εργαζόμενους ε, ε, σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στους οποίους θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου γιατί ε, διακινδυνεύουν